που διακόπησε στις 10 Σεπτεμβρίου 2015 τα συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στις 19 του διατίθενται. Έχετε αντιρρήσεις, ενστάσεις από αυτόν.